Hello everyone. Good evening. Γεια σας λέει Πρόεδρος. Καλησπέρα. Καθίστε για να αρχίσουμε την απόψινή συνεδρίαση. Δεν έχει μπάλα απόψε, οπότε μπορούμε να δουλέψουμε ήρεμα. Πρόκειται για έκτακτη συνεδρία. Έχετε λάβει την μέση διάταξη. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, τότε θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Ανακοινώσει. Έχουμε μία δημόσια ακρόαση που οργανώνει η Επιτροπή Αναφορών σε συνεργασία με την δική μα όσον αφορά τι επιπτώσει των ενδοκρινικών διαταρακτών όσον αφορά τη δημοσιογεία και το περιβάλλον και πώ θα προσαρμόσουμε το ευρωπαϊκό ενωσιακό τέλο πάντων πλαίσιο για την νομοθεσία σε σχέση με τι αμφιβολίες που έχουν υποβληθεί. Αυτό θα γίνει 5η 22 Τρίτου από τι 10 παρατέταρτο στην αίθουσα Γιάν 6Q2. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Έχουμε τώρα κάποιε αλλαγέ όσον αφορά την γραμματεία μα και αυτό έγινε λόγω τη συγκρότηση τη ειδική ερευνητική επιτροπή. ΠΕΣΤ. Η Κριστίνα Μάρμουρ και η Νόρα Χαν Κάπερ πρόκειται να εργαστούν σε εκείνη την ε, ειδική επιτροπή από σήμερα ως ε, αντίστοιχα επικεφαλής γραμματείας και ως ε, διοικητικός υπάλληλος να τους ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία και να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα και βέβαια καλώς να επιστρέψουν όταν ολοκληρωθεί η εγγύη αποστολή τους για σήμερα. Έχουμε διερμηνία σε 16 γλώσσες και ό συνήθως ηλεκτρονικά μπορείτε να βρείτε τα έγγραφα και επίσης μεταδίδεται η συνεδρίασή μας στο ίντερνετ. Επίσης τώρα να εγκρίνουμε τα πρακτικά της 7ης του 2017 και αν δεν έχετε υποβάλει αντιρρησιμότητα του συνεδρίασης τότε θεωρώ ότι εγκρίνονται και προχωρούμε τώρα στο κυρίως πιάτο για απόψε που είναι... Α, όχι, όχι, όχι, όχι, μισό το δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό το κυρίως πιάτο. I have something as a plus here. Um, so we had some um, uh, trilogues going on. Έχουμε κάποιους τριμμένους διαλόγους οι οποίους έχουν την εξελίξη και πρέπει να σας ενημερώσω για το εξής. Έχουμε για τα κτηνιατρικά προϊόντα έναν τριμμένο διάλογο και ο δεύτερος τέτοιος δεύτερος για είναι 26 Δευτέρου. Οπότε και θα συζητηθούν τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία ακόμα εκκρεμούν. Υπήρχαν κάποιες διαφορές ε, και τελευταία φορά ήταν επικοδομητικό το κλίμα και θα δούμε τι άλλα ζητήματα θα πρέπει σε τεχνικό επίπεδο πριν από το, την τρίτη συνάντηση να διεκπληρωθούν Γιατί η τρίτη συνάντηση θα γίνει 22 Τρίτου επίσης. Έχουμε και την έκθεση Τζόφολη που αφορά τις εκθέσεις και την παρακολούθηση σε σχέση με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος και την ε, κατανάλωση καυσίμων των νέων ε, βαρέων φορτηγών και οχημάτων. Θετικό ήταν το κλίμα και εκεί και αυτό σημαίνει ότι οι συνομοθέτες είχαν παρόμοια προσέγγιση για διάφορα σημεία. Οπότε και συμφωνήσαμε όλα τα ζητήματα να εξεταστούν σε τεχνικό επίπεδο και μετά να ξανασυζητηθούν στη δεύτερη συνάντηση της 26ης Μαρτίου. Και τώρα πάμε στο βασικό μας θέμα που είναι η, η έκθεση απολογιστική όσον αφορά την ερευνητική των πραγμάτων επιτροπής του Άμστερνταμ σε σχέση με την μετεγκατάσταση, μετακόμιση τέλο πάντων τη έδρα τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων. Αυτό έγινε 22 Δευτέρου ενεστώ το και επικεφαλής ήταν ο συνέδελφος Τζοβάνι Λαβία. Οπότε ευθύς αμέσως θα πάρει την σκητάλη για να μας τα πει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σας πω σύντομα το τι έγινε σε εκείνη μας την αποστολή στο Άμστερνταμ πάρα πολύ χρήσιμη τόσο ώστε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης όσον αφορά εκεί ε, τα πράγματα για να μπορέσουμε στη συνέχεια να μπορέσουμε να αποφασίσουμε με περισσότερη βεβαιότητα το τι θα γίνει όσον αφορά ε, την ε, μετεγκατάσταση, την μετακόμιση της ε, ΕΜΕ και βεβαίω θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ολλανδική κυβέρνηση διότι μας φιλοξένησε και μας παρέσχε πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την απόφαση και αυτό αφορούσε το, το, τον τόπο εκεί της μετεγκατάστασης και έτσι μπορέσαμε να λύσουμε κάποια ερωτηματικά μια που ήταν πάρα πολύ έντονο το κλίμα στην επίσκεψη, γιατί όλα γίνανε μέσα σε μια μέρα. Και ήδη είχαμε όμως πάρει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Πρώτα-πρώτα, είχαμε πει ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια σημεία όσον αφορά τις σχετικές διαδικασίες από πλευρά Συμβουλίου, που δεν είναι ε, μια διαδικασία που ακολουθείτε συνήθως. Και ε, όλα αυτά είχαν ζητηθεί στα πλαίσια της δουλειάς της ΑΦΚΟ. Πάντως έτσι μπορέσαμε να δούμε ε, τι θα γίνει με την προσωρινή έδρα της ε, ΕΜΑ σύμφωνα με τα όσα πρότεινε η Ολλανδία. Είπαμε ότι εδώ είναι τα πράγματα τεχνολογικά προηγμένα, αλλά χρειάζονται κάποια έργα και δεν θα υπάρξει ιδιαίτερη δυσκολία όλα αυτά να γίνουν. Και όλα αυτά θα γίνουν ε, εμπρόθεσμα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα της μετακόμισης. Οπότε και αυτή η διαδικασία προβλέπεται να ξεκινήσει την πρώτη, πρώτου του 19. Θα ολοκληρωθεί δε μέχρι τέλη Μαρτίου του ιδίου έτους. Αυτό όσον αφορά την προσωρινή έδρα του οργανισμού επίσης μπορέσαμε να εξετάσουμε όλη αυτή την ε, ημέρα τη ισχύ σε συνεργασία με τον εκτελεστικό διευθυντή και έτσι είπαμε ότι θα πρέπει να καταλήξουμε στο ότι δεν θα πρέπει η υπηρεσία να έχει κάποια προβλήματα τα οποία να έχουν σχέση με αυτό το είδος την διπλή μετακόμιση. Δηλαδή πρώτα στην προσωρινή έδρα και μετά στην οριστική. Θα πρέπει ενώ τα πράγματα να γίνουν ε, εύρυθμα τέλο πάντων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και άρα κάποιες διαδικασίες θα πρέπει να γίνουν έστω και πιο αργά εάν θέλουμε ε, μέσα Νοεμβρίου του 2019 να έχει ολοκληρωθεί ή τουλάχιστον να ξεκινήσει η οριστική μετακόμιση. Αυτά όσον αφορά την οριστική έδρα του οργανισμού, η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχει απλώς ο χώρος τον οποίο επισκεφθήκαμε και εκεί θα πρέπει από το α, από το 0 να αρχίσει η ανοικοδόμηση του σχετικού κτηρίου. Και αυτό όμω είναι ένα πρόβλημα, μια πρόκληση για την κυβέρνηση της χώρας, αλλά δεν μας παρέσχουν πάσα διαβεβαίωση και εμείς βέβαια πρόκειται προσεκτικά να ε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αν δούμε ότι ε, αν υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις δεν θα υπάρχει αυτό που λέμε business continuity. Θα πρέπει αυτό να αποφευχθεί πάση θυσία Μα μιλάμε για μια υπηρεσία που θα εξυπηρετεί την υγεία των Ευρωπαίων. Οπότε γι' αυτό και πασχίσαμε σε συνεργασία με τους κοιόδες συζητητές να αποσπάσουμε κάποιες δεσμεύσεις ε, υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία μας δώσανε κατά την επίσκεψη εκεί. Οπότε, η σχετική έκθεση καλύπτει στις λεπτομέρειές της όλα αυτά τα οποία ε, συζητήσαμε έχουμε εκεί όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας τις απαντήσεις από πλευράς Ολλανδών οπότε και εν κατακλείδη θα πρέπει να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τους Ολλανδούς και ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λαβία για την έκθεσή σας νομίζω ότι περιλαμβάνει πολύ σημαντικά στοιχεία για την Επιτροπή μας προκειμένου να προχωρήσουμε και στη ψηφοφορία που έχουμε αργότερα σήμερα. Η αποστολή αυτή αποτελούνταν και από πολλούς άλλους συναδέλφους, τον κύριο Μπόρτσα, τον κύριο Κρούπα, Ρίζ Άλκαν και τον κύριο Πεντιτσίνα και θα ήθελα να τους ρωτήσω αν θέλει κάποιος από τους συμμετέχοντες στην αποστολή να ε, πάρει το λόγο. Αν όχι, να ρωτήσω αν άλλα μέλη της Επιτροπής θα ήθελαν το λόγο. Η κυρία Γκαρντίνη. Να προσθέσω για να έχουμε πιο πλήρη εικόνα ότι ο διευθυντής Ράζη είπε ότι κάποιες δραστηριότητε θα πρέπει να ανασταλούν όπως η κατάρτιση εκπαίδευση γιατί ε, θα υπάρξει κάποια, κάποιο φρενάζ των δραστηριοτήτων γιατί μιλάμε για 14.000 τετραγωνικά ε, μέτρα ε, τα οποία φιλοξενούν τα 27.000 που τώρα έχουν άρα δεν, θα μπορέσει να ανταποκριθεί η υπηρεσία εκτός και όλα γίνουν εμπρόθεσμα επομένως για να μπορέσουμε να τα ολοκληρώσουμε όλα σε αυτό το οκτάμινο ε, θα έχουμε αυτές τις λιγότερες δραστηριότητες αλλά να μην διαθέσουμε ούτε μια μέρα παραπάνω. Βέβαια, μας δώσανε προφορικές ε, διαβεβαιώσεις, δεν έχουμε φυσικά καμιά χειροπιαστή απόδειξη ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Και εγώ λοιπόν αυτό προσδοκώ πάντως αυτό ήταν και αντικείμενο δημοσίευσεων σε εφημερίδες. Ότι δηλαδή μόνο μία εταιρεία ε, απομένει ούτω ώστε να κάνει τα υπόλοιπα για το κτίριο γιατί υπήρχε μια άλλη εταιρεία η οποία αποσύρθηκε από την ε, σύμβαση ε, άλλη παραχωρησίου εταιρεία. Επομένως όλα αυτά μέχρι να σημαίνει λόγια η ΕΜΕ eh, ah, e e θα πάει στο Άμστερνταμ και συνεχίζει αυτή η υπόθεση να μας προβληματίζει. Καλά είναι και το θέμα βέβαια το τι, τι θα γίνει το ρόλο του Κοινοβουλίου, αλλά είναι και το ζήτημα του ότι ο Φάγγελος τον οποίο υπέβαλε στο Συμβούλιο η Ολλανδία δεν είχε πάρα πολύ διάφανος. Τέλος πάντων πήγαμε εκεί πέρα, ε, να κάνουμε τα πράγματα εμείς με, με διαφάνεια και είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα σχετικά έγγραφα αυτά τα οποία χρειάζονται να μας ε, δώσουν για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε οριστικά. Και ήταν επίσης παράλογο το ότι ε, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι είχαμε στην αρχή δύο εταιρείε που είχαν ε, λάβει μέρο στην παραχώρηση του έργου. Αλλά η μία αποσύρθηκε γιατί θεώρησε ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ στριμωγμένο. Άρα εδώ ε, έχουμε χτυπήματα κάτω από τη μέση και θα πρέπει να δούμε το ότι και στο κείμενο μας φαίνεται από τις πρωτο, τροπολογίες ότι τα πράγματα είναι γελία. Θα έπρεπε να φρενάρουμε την όλη υπόθεση και να ερευνήσουμε και να δούμε ποια είναι τα σημεία, τι ξέρουν οι Ολλανδοί που δεν τα αποκαλύπτουν. Να κάνουμε έρευνα και να δούμε κατά πόσον ήταν σύνομη η απόφαση επιλογής της έδρας Ήδη ξέρετε ότι η πόλη του Μιλάνου και το κράτος της Ιταλίας έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γκροστέτ. Όλα αυτά είναι θλιβερά, λέει η κυρία Νομίζω ότι τίθεται να αμφιβόλο η πραγματοποιηθήσα επιλογή. Και παρά τις αμφιβολίες μας τώρα θέτουμε να τα συμφωνηθέντα, τα πράγματα είναι θλιβερά έτσι όπως τώρα εξελίσσονται γιατί είπαμε ότι σε ένα χρόνο θα έχει ε, ολοκληρωθεί η κατάσταση η μετα, μετακόμιση τέλο πάντων και σε ένα χρόνο θα έχει αποχωρήσει το νούμερο βασίλειο επομένως επήγει, επήγει. και δεν μιλάμε τώρα για μια οποιαδήποτε κοινωτική υπηρεσία. Πρόκειται για κάποια υπηρεσία που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο όσον αφορά την επιμέλεια, την προστασία της δημόσιας υγείας. Πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Και η ΕΜΕ δίνει τις ε, εγκρίσεις για θέσεις εμπορία διαφόρων ε, φαρμάκων κλπ. Επίσης και κάποιους πολύ σημαντικούς ελέγχους. Επομένως θα πρέπει να έχει αυτή η υπηρεσία την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη, την καλύτερη δυνατή, ούτω ώστε να μπορούμε να είμαστε συγκρίσιμοι και διαγωνιστικοί με αυτά που γίνονται στη ΣΥΠΑ και αλλού. Άρα όλες αυτές οι αμφιβολίες, τα ερωτηματικά, τι κάνουνε, οδηγούν στο όλοι οι ειδικοί, οι απαραίτητοι πυρογνώμες να σηκώνονται να φεύγουν για να βγαίνουν αλλού που έχουν περισσότερη βεβαιότητα. Ε, άρα, ε, τι θα, θα, θα καταλήξουν να λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις στην υπηρεσία χωρίς αυτό να λαμβάνουν τα πγκέκους που το κάνουν αυτό με τα λογνώση και αυτό είναι ακόμα χειρότερο από όλα τα θέματα στα οποία πάσχει η απόφαση. Και άρα θα πρέπει σήμερα να μπορέσουμε να ασκήσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη πίεση στην ε, κυβέρνηση των κάτω χωρών. Γιατί αυτή 100% είναι υπεύθυνη της απόφασης που διατυπώθηκε και όσον αφορά τις τελικά δημορφωτές επιλογές. Πίεση, πίεση να ασκήσουμε και η ουραδική κυβέρνηση να μετέλθει ό,τι μέσον μπορεί, ούτω ώστε να γίνουν όλα με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, τους ειδικού, τους υπάλληλου, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, αυτοί, αυτοί πρέπει να τα πάνε σε σχολείο, να πάνε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, ή ε, ας κάτσουν να λογαριάσουν και τα ανθρώπινα προβλήματα. Άρα είναι καθήκον μας κυρία Πρόεδρε, επιτακτικό καθήκον να πιέσουμε, να πιέζουμε συνεχώς τους Ολλανδούς ούτω ώστε. Καλά τέλο πάντων δυστυχώ επελέγει το Άμστερνταμ. Οπότε θα πρέπει να δείξει η Ολλανδία ότι τελικά η επιλογή δεν είναι και τόσο κακή. Ευχαριστώ κύριο Μπέναν. Ευχαριστώ. Μια πρόταση να κάνω. Προφανώ από Βρετανό. Άρα δεν θα σα αρέσει και πολύ. Παρ' όλα αυτά, πριν από λίγο καιρό στην Επιτροπή μας ψηφίσαμε ε, στην Επιτροπή μας την αλλαγή χρήσης στη δασοκομεία και ένα, μία από τις διατάξεις ήταν ε, να δοθούν κίνητρα σε ε, προϊόντα μακράς διαρκείας από ξυλία. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους προϊόντα αντί για τσιμέντο και ατσάλι Μήπως θα μπορούσαν ε, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν προκάτ ε, κτίσματα προκειμένου να στεγάσουν ε, τον οργανισμό αυτόν. Θα αρέσει και στους Σκανδιναβούς αυτό. Και ε, φυσικά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι πολύ πιο... Ε, θα, θα ενίσχυε την, ε, την ασφάλεια, την υγεία και θα ήταν και πολύ ωραίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμό Φαρμάκων να στεγάζεται από εδώ και πέρα σε ένα εξαιρετικό και πολύ φιλικό προς το περιβάλλον και την υγεία κτίριο. Ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι θα τύχει μεγάλη υποστήριξη η πρότασή σα, λέει η Πρόεδρο. Αυτά ω προ τον κατάλογο μιλητών. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο άλλο. κύριε Λαβία, θέλετε να επανέλθετε, ε, να σχολιάσετε αυτά που υπόθηκαν. Όχι. Οπότε ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό. Α, κύριε Λαβία, θέλετε το λόγο. Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε, προσπαθήσαμε να ζυγίσουμε, να ισορροπήσουμε τις επιμέρους θέσεις ε, και απόψεις όπως αυτές ε, αναδείχτηκαν στην Επιτροπή και ακόμα και σε αυτό το επίπεδο είχαμε κάποια θέματα και κάποιες κόκκινες γραμμές θεσμικού χαρακτήρα γιατί δεν ήταν δυνατόν να γίνεται έτσι αυτό, να γίνει αυτό έτσι και στο μέλλον από πλευρά απόφαση του Συμβουλίου. Τρόπο απόφαση Συμβουλίου έχει μεγάλη θεσμική συμφωνία και αυτά λέμε στην ε, έκθεση και αυτό ήταν κάτι για το οποίο σημαίνει όλε τι επιτέρυγε του Κοινοβουλίου. Statement. Ε, κάτι σαν δήλωση ε, που αφορά την ψηφοφορία της Επιτροπής μας και τονίζουμε και τα θεσμικά προβλήματα και όσον αφορά αυτά που είπε η κυρία Γκαρντίνη, αυτό που είπε ο κύριο Γκοστέκη, όσα είπε ο Καπούτο, όλα αυτά τα καλύπτουμε, τα καλύπτουμε με τις τροπολογίες τις συμβιβαστικέ. διότι αναγνωρίζουμε τι δυσκολίε. Το υπάρχουν πάρα πολλά σκοτεινά σημεία στην σε διαδικασία. Αποφάσισε μόνο του το Συμβούλιο. Μας άφησε απ' έξω. Άρα, να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα. Θα πρέπει να περισσοθεί την business continuity. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λαβία. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Περνάμε στην πληροφορία. Ελπίζω να έχετε πάρει μαζί σας τις κάρτες σας. Να τις χρησιμοποιήσετε λοιπόν. Έχουμε την κυρία Αγιούσο, η οποία ξέχασε την κάρτα της. Εντάξει, θα ψηφίσετε διανατάσσεως ισχυρός. Και η κυρία Κιλάνεν το ίδιο. Εντάξει. Θα σημειώνουμε τι ψηφίζετε λοιπόν. Περνάμε για την, στην ψηφοφορία για την συναπόφαση, για τις προτάσεις κανονισμού, για την τροποποίηση του παλαιού ε, κανονισμού όσον αφορά την έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, Φαρμάκων. Η συγκητή είναι ο κύριο Λαβία. Ξεκινάμε με, την, με 3 και 4. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και περνάμε στη συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 και 51 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 6 υπέρ, όχι, συγγνώμη, καταπίπτει. Ζητώ συγγνώμη. Περνάμε στην τροπολογία 43. 43. Υπέρ. Όχι, φαίνεται ότι και η 42 καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η 51 από κοινού μαζί με την 50. Οπότε περνάμε στην 43. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αύκο 4. Υπέρ, κατά, δεν είδα. Ξανά. Αύκο 4 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. And it's closed. Πέρας ψηφοφορίας. Αρνητική ψήφος από την κυρία Γιούσο. Θετική ψήφος. Επομένως απορρίπτεται. Αύκο 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη οι επόμενε μάλλον καταπίπτουν, επομένω περνάμε στη συμβαστική τοπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 19 με προφορική τροποποίηση που αντικαθιστά τη λέξη may με το will. Είστε κατά της προφορικής τροπολογίας, όχι τότε μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι παρακάτω τροπολογίες καταπίπτουν και περνάμε στην 23 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είπα 22. Αλλά καταψηφίζετε από ό,τι βλέπω. Θέλετε να ξαναψηφίσουμε για την 22. Όχι, απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην 23. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 και 26 μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 27 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται και περνάμε στην ψηφοφορία επί της ε, έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικά θα γίνει ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. And the vote is... Και η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε και εγκρίνεται. Περνάμε στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος στο σύνολό του, ηλεκτρονικά και πάλι, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση Πέρασε και εγκρίνεται επίσης. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια για την έκθεση. Και έτσι ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας για σήμερα το βράδυ. Θα τα ξαναπούμε στις 14 Μαρτίου σε άλλη μία έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής μας. Τετάρτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Thank you very much. Thank you very much.